So, dear colleagues, please take your seat. It's, it's a little past nine. Έχει. Περάσει, είναι 9 και 3 λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα είναι η στήριξη για τη Μολδαβία. Και θα δώσω τον λόγο αμέσως τον συνάδελφο τον κύριο Σορίν Μόησα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περάσω κατευθείαν στο θέμα. Καλημέρα σε όλους. Λίγα λόγια. Πρώτα, εν ώψη των προκατακτικών συζητήσεων που είχα με συναδέλφους στην ΙΤΑ και στις άλλες επιτροπές ε, εξωτερικών και προπολογισμού για το θέμα αυτό να σας υπενθυμίσω την φύση του μέσω αυτού μιλάμε για μακροοικονομική ενίσχυση τύπου ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ με στόχο το ισοζύγιο πληρωμών και συνήθως συνδέεται με όρους ε, οικονομικής διακυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέρος του ευρύτερου παζλ και υπάρχει αυτή η αιρεσιμότητα που θα οδηγήσει σε μεταρρυθμίσει στην Μολδαβία. Δεν βασίζεται λοιπόν σε έργα, είναι μακροοικονομική βοήθεια, δεν πηγαίνει σε συγκεκριμένα έργα. Ένα τέτοιο πακέτο όμως ε, διαμορφώνεται και η Κομισιόν ε, και η DG ε, την οποία ευχαριστώ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί μου και τους άλλους ηγητές. Μας έχει δώσει ένα non-paper το οποίο παρουσιάζει τις προθέσεις της Κομισιόν και το πώς θα διαπραγματευτούν με τις αρχές της Μολδαβίας και με χαρά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι περιέχει σημαντικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Καταπολέμηση της διαφθοράς, ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, ξέπλυμα χρήματο, δημόσια διοίκηση και βεβαίως ε, τις ε, μεταρρυθμίσει ε, που είπαμε. Όλα αυτά θα έχουν έναν συστημικό αντίκτυπο, ο οποίος οπωσδήποτε θα περιορίσει την δύναμη των ολιγαρχών κτλ. Αυτό είναι μια ενισχύα που έθεσαν οι συνάδελφοι και άλλοι. Να έλαβα μια επιστολή από τον Επίτροπο Μοσκοβισή για το τι πρέπει να γίνει και η αξιολόγηση των όρων επιβεβαιώνει ο Επίτροπος Μοσκοβισή θα είναι αυστηρή. Οπότε οποιαδήποτε ανησυχία ότι θα πετάμε λεφτά σε μια μαύρη τρύπα χωρίς ε, τους ε, σωστούς όρους ε, δεν στέκουν. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι το εάν σεβόμαστε ή όχι το συμφωνημένο πλαίσιο που έχουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χορήγηση της μακροοικονομικής βοήθειας κάτι ανάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα από το 2013 και ε, ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο ήταν δική μας πρωτοβουλία και εδώ και λίγα χρόνια δεν υπήρχε χρηματοδοτική συνδρομή όταν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Προσπαθούμε λοιπόν να πω ότι προσπαθούμε τώρα να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Θα έχουμε μια καθυστέρηση και διαπραγματεύσει με τα άλλα θεσμικά οργάνα μέχρι να έχουμε το σωστό πλαίσιο και οι επιπλέον εγγύησει που λάβαμε από την Κομισιόν και αυτές τις θέλουμε και δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς μέχρι τότε να στείλουμε την βοήθεια αυτή στην Μολδαβία και θα είναι ένα λάθος μήνυμα για τη Μολδαβία και τους άλλους εταίρους. Επίσης αν γίνει κάτι τέτοιο θα χάσουμε και οποιοδήποτε μέσο πίεσης για τις μεταρρυθμίσεις. Στην επιστολή που ανέφερα λοιπόν το δικαίωμα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρο και το εγγυάται ο Επίτροπο Μοσκοβισή θα λάβει την ίδια πληροφόρηση ταυτόχρονα με την Επιτροπή του, των Καρτών Μπελών και το Συμβουλίο. Και οι υπηρεσίε μας θα συνεργαστούν για να βρουν ακριβώ τις λεπτομέρειες. Η λύση λοιπόν είναι ένα πακέτο αίρεσιμότητα που υπάρχει, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται και θα δεχτεί νομίζω η Μολδαβία, μα το έχουν πει, και θα υπάρξει γενικώ μια μεταρρύθμιση σεβόμενη πάντα τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο προτάσει λοιπόν που έχω να κάνω στου συναδέλφου. όταν θα σκεφτούν τι τροπολογίε του. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να εκφράσουμε ανησυχίες στα εκτιμώντας της απόφασης για να δοθεί κατεύθυνση στην Κομισιόν και ελπίζω σε αντίθεση με κάποιες από τις ε, τροπολογίες στην ΑΦΕΤ να έχουμε κάποιους όρους οι οποίοι δεν θα είναι αδύνατον να εκπληρωθούν κάποιες από τις τροπολογίες στην ΑΦΕΤ ε, θέλουν η Μολδαβία να είναι ε, καλύτερη από τη Γερμανία μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, κάτι το οποίο μάλλον δεν γίνεται. Οπότε καλό είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Μολδαβία και το κάνουμε σοβαρά, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές για το τι μπορεί να επιτευχθεί. Αλλιώς, ξέρετε, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. δεν θα τους βοηθήσουμε τελικά. Οπότε ε, βεβαίως ρεαλιστές δεν σημαίνει ότι παριστάνουμε ότι θέτουμε όρους. Χρειάζονται όροι και όπως είπα αυτά έχουν συστημικές συνέπειες και οι Μολδαβοί είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να δεχτούν κάτι τέτοιο αλλά πρέπει να έχουμε όρους οι οποίοι ρεαλιστικά να μπορούν να εκπληρωθούν έχοντας όλα αυτά κατά νου Αναμένω τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Η προθεσμία είναι μέχρι την 1η Απριλίου. Έχουν λοιπόν όλοι καιρό να το σκεφτούν. Και αναμένω και την συνεργασία μαζί σας για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω στην ψηφοφορία του Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στους για το έλκο κύριος Βίγκλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα, κύριε Πρεσβευτά. Ευχαριστούμε για την βαθιά και διεξοδική και πολύ εντελεχή δουλειά του συναδέλφου εισηγητή για το θέμα αυτό. Και εγώ να εκφράσω τη σκέψη ότι καλώς λειτουργεί με διαφανή τρόπο η Επιτροπή και έχουμε το non-paper για να κατανοήσουμε ακριβώ ποιε είναι οι προθέσει τη. Είναι σημαντικό. Διότι το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί με την απόλυτα διαφανή και σαφή και ξεκάθαρη ρησιμότητα που, χρειάζεται, ε, που χρειάζεται για, για να δούμε τι προθέσει τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Όσο ήθιστε σε αυτή την Επιτροπή, θέλω να είμαι ειλικρινή και έντιμο και να εκφράσω την απογοήτευσή μα ω προ τι εξελίξει στην Μολδαβία. Αυτό αληθεύει και για την οικονομία και το εμπόριο. Είμαστε αρκετά δυσαρεστημένοι. Τέλο πάντων, να πω ότι δεν αισθανόμαστε άνετα με τον ε, βαθμό ε, ε έγκριση που δίνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπόριο και την οικονομία τη Μολδαβία. Οι δυνατότητε αυτέ είχαν προσφερθεί και με την αρχική υποστήριξη της Επιτροπής μα της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου, στην προηγούμενη θητεία κιόλα. Την περασμένη δεκαετία, αν θυμάμαι καλά. Οι δυνατότητες αυτές ήταν σημαντικές. Τότε. Συμφωνώ λοιπόν κατά μεγάλο μέρος με το να αλλάξουν ε, τα κριτήρια για την μακροοικονομική βοήθεια και να αλλάξουν και οι δόσεις, βλέποντας το βαθμό εκπλήρωσης των στόχων της Μολδαβίας και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει, τις προθεσμίες και πρέπει να είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας να εξακολουθήσει η στήριξη της δημοκρατίας της Μολδαβίας μεν, για να είμαστε παρόντες εκεί όταν χρειάζεται και να επιβεβαιώσουμε την ε, πάγια στάση μας ότι είμαστε η ένωση που θέλει να σταθεί δίπλα τους και όχι απλώς ότι βασίζομαστε σε συμφέροντα και την εξυπηρέτησή τους, αλλά νομίζω μεταξύ των ε, εταίρων μας προς Ανατολές τα πράγματα του χρόνου θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, όχι πιο απλά. Θα πρέπει λοιπόν η δεσμευσή μα προ τη Μολδαβία στα πλαίσια αυτή τη Επιτροπή ΙΝΤΑ να διατηρηθεί. Ευχαριστούμε για την Άλντε, ο κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μολδαβία είναι σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Και η συμφωνία μα είναι μια ένδειξη τη καλή σχέση συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μολδαβία. Για την ε, καλή εφαρμογή τη ει και και συνεισφαιρική συμφωνία, για την οικονομία και το εμπόριο, τι μεταρρυθμίσει που χρειάζονται, θα πρέπει να υπάρξει υλοποίηση στην πράξη, στην Μολδαβία. Επίση, η τραπεζική κρίση στη Μολδαβία ήταν κρίσιμη σημασία. Η εποπτεία του κλάδου αυτού δεν ήταν επαρκής, ενώ με την κρίση δυσκόλυψε η πρόσβαση στα δάνεια και αυξήθηκε το κόστος τους. Η πολιτική κρίση και η απουσία σταθερής και ανεμπόδιστης προσπάθειας μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση καθιστά πολύ δύσκολη την υλοποίηση στην πράξη, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Επίσης η πολιτικοποίηση και η ε, δυσκολία της ανεμπόδιστης δουλειάς των αριθμιστικών φορέων σε τομείς όπως η ενέργεια, το εμπόριο και οι δημόσιες προμήθειες δημιουργούν ανησυχίες και αντίκενται στις αρχές της ε, εισβάθους και σφαιρικής συμφωνίας. Είναι λοιπόν αρκετές προκλήσεις που προκύπτουν εδώ. Η ιδεοντολογία και η ακαιρεότητα είναι σημαντικά στοιχεία στα πολιτικά πράγματα. Πρέπει να ενισχυθεί το πολιτικό σύστημα τη χώρα, καθώ επηρεάζει και τι ροέ τη άμεση ε, ξένη βοήθεια και των επενδύσεων. Ε, το κράτο δικαίου πρέπει να γίνεται σεβαστό και να υπάρχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για τι ξένε επενδύσει. Όλα αυτά τα ζητήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να υποστηριχθεί η Μολδαβία στην πορεία αυτή τη ανάπτυξή τη με προσφορά μακροοικονομική βοήθεια που είναι ένα μόνο τρόπο για να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στήριξή τη. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται συστηματικά για όλε τι μελλοντικέ εξελίξει στην Μολδαβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάκουλα. Για την ΓΟΕ ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ και τον συγγητή για τη δουλειά που έχει κάνει που πηγαίνει προς την κατεύθυνση ότι η κατάσταση στην Πολταβία ε, απαιτεί ακόμα πολλές βελτιώσεις ειδικά όσον αφορά τη δημοκρατία, το κρατός δικαίου και τα λοιπά. Θα ήθελα όμως να συμφωνήσω με τον εισηγητή λέγοντας δηλαδή ότι όταν αποφασίζουμε για τέτοια πράγματα πρέπει να έχουμε κατά νου το εξής. Πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη της χώρας για να μπορεί από μόνη τη να δει πώς θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις, πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα συμφέροντα του λαού της ε, χώρας. η ανάπτυξη της γεωργίας, ε, της συνοποιίας κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω ταυτόχρονα. Ε, ήθελα να πω το εξής πρέπει να είναι πιο σαφής η όρη. Βλέποντας την ε, σχέση με την συνεδρίαση την απόψινή με τον Επίτροπο Χάν στην Άφετη για το στρατηγικό διάλογο με τις ε, χώρες της, δυτικής, της ανατολικής γειτονίας. Χρειάζεται κάποια αυστηρότητα. Για να υπάρξει ε, Βλέπουμε εδώ πέρα μία μείωση των κονδυλίων ε, στην Μολδαβία όπως προτείνει η Κομισιόν. Μα ε, τότε πώς θα έχουμε πιστώσεις, πώς θα έχουμε άμεση στήριξη ε, χρημάτων τα οποία δεν θα ε, ρέουν ξανά πίσω στον προπολογισμό της κοινότητας. Ε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπως αυστηροί, να δούμε τι κάνουμε στον νέο τομέα, τι κάνουμε στον άλλον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Τελικά το θέμα πρέπει να είναι πολιτικές διαδικασίες στη χώρα, η, αξε, η ανεξαρτησία της ε, τυπικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα πολύ εξαρτημένης, όλα αυτά να βοηθηθούν με την δική μας τη βοήθεια, να συνεισφέρουμε στην εξυγίανση της χώρας. Σας ευχαριστώ πράσινοι και οι FTD δεν είναι εδώ, είναι πολύ νωρί για να ξυπνήσουν. Δίνω λοιπόν το λόγο πρώτα στην Κομισιόν και μετά στην Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η Μολδαβία από το 2014, τα τέλη του 2014, αντιμετωπίζει μια δύσκολη μακροοικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. Έχει υποστεί διάφορα σοκ στην οικονομία της, τραπεζική κρίση, εν μέρη λόγω τραπεζικής απάτης μεγάλης κλίμακας, ύφεση, ε, προβλήματα με τους εταίρους της, δηλαδή τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία έχει μειωθεί η στήριξη των βασικών δωρητών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι προβλήματα που μαστίζουν την οικονομία της Μορδαβίας. Και Όλα αυτά υπάρχουν μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση που να κάνει τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Ο Πρωθυπουργό Φιλίπ στα 2016 έφτασε στην εξουσία και διορίστηκε κεντρικός τραπεζίτης, επίσης υπέρμαχος των μεταρρυθμίσεων που προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση μαζί με τον ε, Διευθυντή της ε, Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμόσει τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Το Φεβρουάριο πέρσι ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα υιοθετήθηκε από τις αρχές, πρόγραμμα μητερρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της ε, δικαιοσύνης, αλλά και πάρα πολλέ οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για να αξιοποιήσουμε αυτό το momentum που υπάρχει τώρα, να, να αξιοποιήσουμε την ορμή για μεταρρυθμίσεις και να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα. Με αιρεσιμότητα βεβαίως, με προαπαιτούμενα, ισχυρά, ε, σε διάφορους τομείς. Βασικό θέμα του προγράμματος είναι η μεταρρύθμιση της διοίκησης, της διακυβέρνησης στο τομέα των τραπεζών, στον ενεργειακό τομέα, ανεξαρτησία ε, του ρυθμιστή της αρχής ρύθμισης ε, ενέργειας, εξωτερικός οικονομικός έλεγχος και διάφορες άλλες μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και ε, με σκοπό την εφαρμογή των δεσμεύσεων βάσει της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όλα αυτές η, συμμετοχή του Δουνουτού πάντοτε υπάρχει όταν ε, τηρούνται μεταρρυθμίσει ε, στον οικονομικό τομέα αλλά και στο δικαστικό τομέα και για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προτείνεται όλα αυτά να συνδεθούν με την πρόοδο και στη διαδικασία σύνδεσης. Κάθε δόση που θα απελευθερώνεται, θα εκταμιεύεται, θα συνδέεται με την θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εμείς έχουμε πρώτα υπεροαπαιτούμενα σε κάθε εκταμίευση δόσης. Συνήθως η πρώτη εκταμίευση του δονοτού γίνεται όταν έχει γίνει ε, σωστή εκκίνηση του προγράμματος. Η Επιτροπή όμως προτείνει να υπάρχει ε, σοβαρή αξιολόγηση, ισχυρή αξιολόγηση και να εκταμιεύεται ε, η δόση κάθε φορά που θα επιτυχάνεται ικανοποιητική αξιολόγηση. Και όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσουμε και με άλλες οικονομικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε λοιπόν οικονομική βοήθεια. Η Μορδαβία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει, ως ενίσχυση, να υπάρξει ενίσχυση βοήθεια με τη, ε, τη μορφή της ενίσχυσης πληρείται δηλαδή ο κατάλογος κριτηρίων του ΔΝΤΑΦ ε, ούσα η πιο φτωχή χώρα στην περιοχή και ούσα η πιο χρεωμένη ε, χώρα. Επομένως γι' αυτό λέμε ότι η βοήθεια πρέπει να δοθεί με, την ε, τη μορφή του grant της ενίσχυσης. Πληρείται ο σχετικός κατάλογος κριτηρίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι σημαντικό ωστόσο και συμφωνώ με τον εισηγητή οι συνομοθέτες, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, αν θέλουν να τροποποιήσουν το κείμενο, να εστιάσουν την προσοχή τους στις αιτιολογικές σκέψεις, για να μην θέσουν σε κίνδυνο το δύσκολο συμβιβασμό στον οποίο έφτασαν πριν από τρία-τέσσερα χρόνια επί τη ευκαιρία της κοινή δήλωση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την οικονομική βοήθεια. Επομένως, καλό θα είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στις αιτιολογικές σκέψεις, όπως λέει και ο εισηγητής, και σε μια επιστολή που εστάλει χθε από τον αρμόδιο Επίτροπο Μοσκοβισή σε απάντηση της επιστολής του εισηγητή κ. Μόισα, αναφέρεται ότι ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτή ενημέρωση για το μνημόνιο της Μολδαβίας, τακτή ενημέρωση και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας της Επιτροπολογίας. Αυτό προβλέπεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει άμεσα να διαβάζονται και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μετά τη δεκταβίευση κάθε δόσης και... και μπορούμε και γραπτός να σας υποβάλουμε όποια στοιχεία ε, επιθυμείτε. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την πρόταση χωρίς σημαντικές τροπολογίες και αν υπάρχουν τροπολογίες να υπάρξουν μόνο για τις αιτιολογικές σκέψεις. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι θα έχουμε πολύ αυστηρούς ελέγχους για την αξιοποίηση του Ταμείου. Έχει γίνει συνολική αξιολόγηση των οικονομικών και διοικητικών κυκλωμάτων. Επιχειρησιακή αξιολόγηση προηγείται κάθε παρέμβαση του ΔΝΤ. Το μνημόνιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρέωση να επιτρέπονται επιθεωρήσεις, να υπάρχει προσφυγή στο ελεγκτικό συνέδριο, να υπάρχουν διατάξεις που θα έχουμε αυτόματη διακοπή εκταμίευσης οποιασδήποτε ε, δόσεις αν ανοιχνευτεί οποιαδήποτε παρατυπία, αλλά και ε, ε, early repayment, να υπάρχει πρόβλεψη να επιβληθεί, να ε, ε, αποπληρωθεί το δάνειο ε, νωρίτερα εάν αυτό απαιτείται. Πρέπει να πούμε ότι η Μολδαβία, όπως και άλλοι που είναι σε πρόγραμμα, έχουν σοβαρά προβλήματα διοίκησης και διακυβέρνησης όμως νομίζουμε ότι έχουμε σταθμίσει σωστά το κίνδυνο για τις χώρες μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρόγραμμα και τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα που έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και ελπίζουμε η Επιτροπή να στηρίξει την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλημέρα η Μολδαβία μετά από μια, πολιτική, μια περίοδο πολιτική αστάθεια την τελευταία χρονιά έχει νέο πρόεδρο. Μόλι επέστρεψε στο δεύτερο ταξίδι του στη Μόσχα ο πρόεδρο αυτό, ο νέο εκλεγμένο, για να βελτιώσει τι σχέσει τη χώρα με την ε, Ομοσπονδία τη Ρωσία. Το ευχόμαστε Καλή τύχη. Ωστόσο, η Δημοκρατία τη Μολδαβία, παρά την φαινομενική πρόσφατη σταθερότητα, έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει, όπω την ε, διαφθορά, την διακυβέρνηση, τα προλογικά, τα δημοσιονομικά, την αδυναμία πληρωμών, την έλλειψη ανάπτυξη και πρέπει διεξοδικά να ερευνήσει την ε, τεράστια τραπεζική απάτη που οδήγησε σε κρίση την, ε, τον κλάδο τη χώρα το 2014 για την οικονομία τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τι εξελίξει αυτέ στενά βάση και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Εξωτερικών του Φεβρουαρίου του 2016 που παραμένουν ακόμη σε ισχύ. Πριν από μία εβδομάδα, στις 13 Μαρτίου, δημοσιεύτηκε έκθεση για τη Μολδαβία που αποτιμά την πρόοδο, πρόοδο για την υλοποίηση της ε, συμφωνίας ε, και το, την ανάγκη των ε, εναπομεινασών μεταρρυθμίσεων. με παρουσία του Πρωθυπουργού ε, Φίλιπ και τη ε, ε, τη εκπροσώπου Μογκερίνη, θα οργανωθεί συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα για να συζητηθούν οι εξελίξει στο επίπεδο των δύο συμφωνιών. Οι εκταμιεύσει βάσει του προγράμματο MFA θα προχωρήσουν υπό την αιγίδα του Διεθνού Νομοσπονδιακού Ταμείου και βεβαίω θα συμφωνηθούν και προποθέσει πολιτική αρεσιμότητα από τι δύο πλευρέ. Όλα αυτά γίνονται σε στενό συντονισμό με τα προγράμματα προσαρμογή και μεταρρυθμίσεων που η Μολδαβία έχει συμφωνήσει και με τη Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα και στο πλαίσιο τη υποστήριξη ε, τη δική μα προ τον προπολογισμό του. Η στήριξη προ τον προπολογισμό έχει παρόμοια αιρεσιμότητα. Ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, καταπολέμηση τη διαφορά, για να αναφέρω μόνο τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία. Πιστεύουμε ότι η Μολδαβία μπόρεσε να κάνει κάποιε σχετικέ μεταρρυθμίσει στου τελευταίου μήνε, αλλά είναι σημαντικό να συνεχιστούν και να εφαρμοστούν χωρί παναχωρήσει. Ελπίζουμε ότι και εσεί θα συμβάλλετε κι άλλο στον συγχρονισμό τη Μολδαβία, όπω τι εμπορικέ ε, συναλλαγέ. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά ώστε η Μολδαβία να δράξει οικονομικέ ευκαιρίες. Με περισσότερε εμπορικέ δυνατότητε και εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντα περισσότερα στου νέου και την εργασιακή και, τους και την ηλικιακή ομάδα των νέων που πρόκειται να εργαστούν. Όπως εκθέσετε στα συμπεράσματα του Φεβρουαρίου του 2016, ε, χρειάζονται χειροπιαστά αποτελέσματα για να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Thanks a lot and hope... Ευχαριστούμε. Όντως ελπίζουμε ότι οι βελτιώσεις αυτές θα ε, γίνουν και πράξη. Με συγχωρείτε, κύριο Σόλτ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την υπηρεσία εξωτερικών. Αναφέρατε τις ε, πρόοδους που έχει πτυχεί η δικαιοσύνη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαδικασίες ε, καθυστερημένες, διαστρεβλωμένες, υπάρχουν άτομα στη φυλακή με τραγικές συνθήκες, με αλυσίδες στα πόδια σε κατοίκον περιορισμό και περνάνε μήνες και τα χρόνια χωρίς να γίνεται τίποτα. Και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου και οι δικηγόροι δηλαδή πλέον έχουν παρετηθεί. Ε, δεν είμαι υπέρ του να παρεμβαίνουμε σε άλλες χώρες, αλλά εδώ πέρα κάτι πρέπει να γίνει. Πώς παρακολουθείτε λοιπόν αυτήν την διαδικασία, κύριε Σίμπελ. Ευχαριστώ. Απαντήστε αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Σε πάμπολες ε, περιστάσει και με την επίσκεψη του Προέδρου τη Χώρα τη Βρυξέλλη, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Και ο πρόεδρο Τούσκ και ο πρόεδρο Γιούνκερ τα ε, επισημάνανε. Υπάρχει πολλή δουλειά που απομένει να γίνει λοιπόν σε σχέση με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο. Το έχουμε τονίσει σε απειράριθμε περιστάσει. οι ε, υποθέσει που αναφέρατε και υπάρχουν και άλλε. Όχι μόνο κατά πολιτικών, αλλά δημοσιογράφων, δικηγόρων. Παρακολουθούνται στενά. Και θέλουμε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πολιτικοποίηση. Είναι ανησυχία που συνεχίζουμε να την εκφράζουμε και σα διαβεβαιώ ότι το Συμβούλιο για να συζητήσει το θέμα της ε, Σχέση συνεργασία θα ε, επιμείνει και σε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστούμε. Και τώρα ο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και σκιώδεις για τις επικοδομητικές τους παρατηρήσεις σήμερα και για την επικοδομητική και ρεαλιστική τους στάση. Αυτό που προτείνω είναι να συναντηθώ προσωπικά με τον καθένα σας την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα πριν, για τη, πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των και βάσει όλων των πληροφοριών που θα συγκεντρώσουμε, των προτεραιοτήτων και των παρατηρήσεων σας, να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε. Και μετά μπορούμε να οργανώσουμε και μια ομαδική συνάντηση με όλους τους σκιώδεις. Πραγματικά όμως θέλω να υπάρξει συνένεση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ή δυνατόν και πριν την ε, καταληκτική προθεσμία για τις τοπολογίες. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τη ρεαλιστική, επιφυλακτική, αλλά παρόλα αυτά επικοδομητική του στάση στο θέμα. Ε, εκεί θα αναζητήσουμε το σωστό σημείο ισορροπία. Θα αγωνιστούμε για να αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόφαση χωρί ή δυνατόν να διαταραχθεί αυτή η τόσο προσεκτικά διαπραγματευμένη συμφωνία. Για να μην περάσουμε σε μια γκρίζα ζώνη βεβαιότητα. Όχι μόνο για αυτό το πακέτο βοήθεια, ενδεχομένω και για μελλοντικά ή άλλα που θα πάνε στι χώρε τη ίδια γειτονιά ή προ Ανατολέ. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτησή μα. 5 Απριλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών το μεσημέρι στι 12 και η ψηφοφορία θα γίνει 3 και 4 Μαΐου. Ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, το σημείο 9 ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη χορήγηση συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στη Σρι Λάγκα. Γενικευμένων προτιμήσεων συν. Η Σρι Λάγκα ζήτησε να της χορηγηθεί αυτό το καθεστώς στις 12 Ιουλίου. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν δίνει προτιμησιακή πρόσβαση σε χώρες που καλύπτουν περίπου το 6% όλων των δασμολογικών γραμμών. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες αυτές πρέπει να δεσμευθούν ότι θα βελτιώσουν και θα επιβάλλουν 27 διεθνείς συμβάσεις. Στις 11 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει μια κατεξοσοδότηση πράξη που θα χορηγήσει το καθεστώς αυτό στη Στριλάνκα. Κατόπιν ετήματος πολλών ε, βουλευτών, αποφασίσαμε να παρατείνουμε το διάστημα για την εξέταση του θέματος αυτού μέχρι τις 11 Μαΐου, ώστε να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. και να ε, αποφανθούμε αν μπορούμε να στηρίξουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλουμε να την απορρίψουμε. Είμαστε εντός προγράμματος και έχουμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε και να συζητήσουμε τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Σιλάνκα. Και θα τα συζητήσουμε σήμερα με εμπειρογνώμονε επί του θέματο. Είναι προφανέ. ότι οι συμβάσεις του 87 και 98 για τα εργασιακά δικαιώματα δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται ακόμα. Πρέπει και αυτό το ζήτημα να συζητηθεί. Σήμερα έχουμε μαζί μας τρεις εμπειρογνώμονες. Θα τους προσκαλέσω να λάβουν το λόγο καθένας τουλάχιστον για πέντε λεπτά. Ώστε να έχουμε και χρόνο για συζήτηση μετά, μεταξύ των βουλευτών. Περίπου 45 λεπτά προβλέπονται για αυτό το θέμα συνολικά. Οπότε μάλλον θα σας περιορίσω, συνάδελφοι, και στο χρόνο ομιλίας σας τελικά. Πρώτα απ' όλα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ε, θα δώσω το λόγο και στην Επιτροπή και στον Πρεσβευτή της Σρι Λάνκας. Ο καθένας για πέντε λεπτά. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Yes, thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω λίγο για το υπόβαθρο, το ιστορικό το 2010 έχασε η Σρι Λάγκα το σύστημα γενικεμένων προστιμήσεων ΣΥΝ λόγω του ε, ανεπαρκών επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λόγω του ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη. Τον Ιανουάριο του 2015 άλλαξε το πολιτικό καθεστώς, είχαμε εκλογή νέου Προέδρου και ο Ρανίλ Πρεμασίγκα έγινε Πρωθυπουργό. Η νέα κυβέρνηση καθόρισε ένα πρόγραμμα βαθέων μεταρρυθμίσεων για να λυθούν τα προβλήματα διακυβέρνησης, διαχείρισης, για να υπάρξει κράτος δικαίου, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, συμφιλίωση και λογοδοσία μετά από τον εμφύλιο πόλεμο. Αναγνωρίζουμε πλήρως την πρόοδο που έχει σημειώσει ενώσει η χώρα αυτή τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει αποκαταστήσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις, είναι εν εξελίξη η σύνταξη νέου συντάγματος που θα οδηγήσει σε πολιτική ρύθμιση, επίλυση των προβλημάτων με εκχώρηση εξουσιών, θα καταργηθεί η εκτελεστική προεδρία και θα υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου, του εκλογικού συστήματος. Έχουν γίνει βήματα για την εθνική συμφιλίωση. Υπάρχει ένας προσωρινός μηχανισμός λογοδοσίας και δικαστικής εξουσίας. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί με το ψήφιο των Εθνών που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 να πράξει τα δέοντα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα κυβέρνηση συνεργάζεται ομαλά, επικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε ξεκινήσει έναν ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο για πολύ λεπτά ζητήματα. Ο Πρωθυπουργό τη Σρι ήταν στι Βρυξέλλε τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Υπουργό Διεθνού Εμπορίου έχει έρθει στι Βρυξέλλε δύο φορέ φέτο και ο Υπουργό Οικονομικών ήρθε στι Βρυξέλλε τον Ιανουάριο του τρέχοντο έτο. Πέρσι φτιάξαμε μια νέα ομάδα εργασία για τη διακυβέρνηση, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Κολόμπο και τα θέματα που συζήτησε η ομάδα εργασίας είναι πολύ πιο ευρεία από τα προαπαιτούμενα για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει πολιτική βούληση να προχωρήσει πολύ περισσότερο από τα ελάχιστα προτα... προαπαιτούμενα για να χέρι του καθεστώτος του συστήματος γενικεμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση πολύ επικοδομητικά με τους ειδικού εισηγητές και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Έχει απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ειδικού εισηγητές και πολλοί από αυτούς επισκέφτηκαν τη χώρα πέρσι. Όπως αναφέρεται στην ολοκληρωμένη ε, έκθεση που δημοσιεύτηκε στις αρχές Μαρτίου για τη Σρι από ε, τον ε, αρμόδιο επίτροπο και είπα το εκπρόσωπο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα υπάρξει νέο ψήφισμα το οποίο θα προσυπογράψει η κυβέρνηση της Σρι και θα δίδονται δύο, δύο χρόνια έξτρα επιπρόσθετα για να μπορέσει η κυβέρνηση να επιτύχει αυτά στα οποία δεσμεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Ο κατάλογος με τις δεσμεύσεις ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος πράγματι, υπερβολικά φιλόδοξος τότε και λογικό είναι που δεν εκπληρώθηκαν όλα. Παρ' όλα αυτά ε, έχει σημειώσει πρόοδο αυτή η χώρα και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί παράταση. Ε, η νέα από κοινού ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Ανώτερων Στελεχών είπα των εκπροσώπων και υψηλών αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών θα οργανωθεί στη χώρα αυτή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έχος. Πράγματι, μερικές φορές γενικά ο ρυθμός είναι πιο αργός από αυτό που ε, θα θέλαμε εμείς. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι όντως δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις αυτές και η κυβέρνηση της Σρι Λάγκα χρειάζεται τη διεθνή στήριξη για να τις φέρει σε πέρας. Ορισμένα στοιχεία στη Σρι Λάγκα και ενδεχομένω στο εξωτερικό προσπαθούν να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία και αυτό πρέπει να υποθεί. Σίγουρα μένουν πολλά να γίνουν, όμω η Σρι Λάγκα είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και η τάση έχει θετικό πρόσημο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ το και εγώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Γκαλίνα ήταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν τη βλέπω. Ποιο εκπροσωπεί την Επιτροπή, εσεί, παρακαλώ. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ. Καλημέρα η κυρία Ανταλίνα που ουσιάζει είναι στην Αργεντινή και πραγματεύεται για την Μερκοσούρ. Βεβαίω θα ήθελε να είναι εδώ την αντικαθιστώ εγώ και ο, είμαι ο Νίκος Ζαΐμης, ε, σύμβουλος του DigiTrade, ε, υπεύθυνο για την βιώσιμη ανάπτυξη και τις γενικευμένες ε, προτιμήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα. Ήδη είχα μία συζήτηση το Δεκέμβριο πέρσι, αλλά αυτή είναι η πρώτη συζήτηση μετά την έγκριση της απόφασης της Κομισιόν για τη χορήγηση γενικευμένου στήματος προτιμήσεων στην Σριλάνκα. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ σύντομα σε κάποια πράγματα. Ε, η προηγούμενη συνάδελφο μίλησε 4 λεπτά και μετά η δευτερόλεπτα. θα μιλήσω λίγο για την διαδικασία την αξιολόγηση και το ευρύτερο πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την διαδικασία, πολλέ από αυτέ τι ε, πληροφορίε υπάρχουν ήδη στο έγγραφο εργασία, ε, στο σχέδιο πράξη κατεξοδότηση. Δεν θα τα επαναλάβω, αλλά τα βασικά στοιχεία που εφάρμοσε η Σρι Λάνκα πέρσι τον Ιούλιο όταν η Κομισιόν έπρεπε να, εξηγεί, να εξετάσει σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό εάν ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλεξιμότητος, τα οποία είναι ε, κριτήρια ευπάθεια οικονομικά, τα οποία ανταποκρίνεται, δεύτερον η κύρωση, χωρίς ε, επιφυλάξεις για τις 27 συμβάσεις ε, του κανονισμού του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων και τέλος δέσμευση να υπάρξει παρακολούθηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έληφθη μια απόφαση στις 11 Ιανουαρίου εντό έξι μηνών μια προθεσμία που ορίζει ο κανονισμός θέλω να υπενθυμίσω είχαμε σχόλια συχνά από τρίτες χώρες όπω θα μπορούσαμε να αναστείλουμε να περιμένουμε κτλ Δυστυχώ αυτό δεν γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό η Κομισιόν πρέπει να λάβει μια απόφαση εντό εξαμήνου Όσον αφορά τώρα την αξιολόγησή μας, η αξιολόγηση περιέχεται στο έγγραφο εργασίας. Ε, το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια σοβαρή μη εφαρμογή των 27 συμβάσεων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, ότι όλα είναι τέλεια στην Σρι Λάνκα. Καθόλου, κάθε άλλο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα έχουμε όπως έχουμε πει πολλές φορές στην Επιτροπή. Είναι ένα θέμα κινήτρων, δεν είναι κάποια ανταμοιβή για χώρε οι οποίες ε, έχουν ήδη επιτύχει κάποια πράγματα. Αλλιώς ε, θα γινόταν μόνο σε χώρε χώρες, ε, Νορβηγία, Ελβετία και ίσως ούτε και σε αυτές. Λοιπόν, η Κομισιόν έχει βρει με τη συνεργασία της Υπηρεσίας εσωτερικής Δράσης και άλλων υπηρεσιών, είχε για την απασχόληση, κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στις διάφορες συμβάσεις ε, και τα οποία βεβαίως θα τα δούμε και στην παρακολούθηση του GSP+. Η ανάλυση της ε, Κομισιόν έχει τρεις πυλώνες ε, όπου βλέπουμε τις συλλήψεις αλλά βλέπουμε και πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά και του περιορισμού που αντιμετωπίζει ο δικαιούχο. Λοιπόν, και στα τρία μέτωπα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Λάγκα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του κανονισμού, Όπω ακριβώ έχουμε λοιπόν εφαρμόσει τον κανονισμό και σε άλλου δικαιούχου. η Κομισιόν αποφάσισε να χορηγήσει το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων και στη Λάγκα. Τώρα λίγα λόγια για το πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις του κανονισμού. Αυτό το σύστημα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του νέου ε, σχήματος. Λοιπόν, στο παρελθόν έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, τα μέσα παρακολούθησης μέσω πίνακα βαθμολογίας, ε, διαλόγου, δεν θα τα επαναλάβω. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημείο που διαφέρει λίγο στην περίπτωση της Σρι ότι η παρακολούθηση αυτή θα ενισχυθεί από δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε εκ παραλίλου την παρακολούθηση της Κομισιόν να δούμε τις δεσμεύσεις της ε, Σρι ε, σε ε, δύο πτυχές. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ανέφερε η συνάδελφος, η διμερής πτυχή ήδη κάνουμε ένα διάλογο για τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου συζητούμε όλα τα ζητήματα που περιέχονται στο GSP+. Βέβαια, ο διάλογο είναι ευρύτερο και άλλα οι ελλείψει, ε, τι οποίε βλέπουμε είναι κομμάτι του διαλόγου ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι η πτυχή του ΟΗΕ και πάλι, όπω και με άλλου δικαιούχου Έχουμε την πτυχή του ΟΗΕ όπου υπάρχει μια έντονη συζήτηση στον ΟΗΕ όπω μόλι ακούσαμε αύριο θα γίνει μια συζήτηση στη Γενέβη στο Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη Σρι Λάνκα και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμφωνία, ότι θα έχουμε ένα νέο ψήφισμα το οποίο θα προβλέπει άλλη μια διετή πιθανότατα περίοδο εντός της οποίας η Σρι Λάνκα θα πρέπει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που περιέχονται στο ψήφισμα. Οπότε δύο πτυχές πέρα από το παρακολούθηση GSP+. Τώρα, θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι οπωσδήποτε ο κανονισμός είναι τώρα ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Υπάρχει μια μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Σρι θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και τη διαδικασία. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, δεχόμενη ή απορρίπτοντας ε, την εφαρμογή αυτή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μερικέ φορέ τα πράγματα δεν είναι απλώ άσπρα ή μαύρα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, υλοποίηση των 27 συμβάσεων. Όχι δηλαδή μόνο να σκεφτούμε αν θα εγκρίνουμε, θα απορρίψουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά μήπω υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα οδικό χάρτη και το καθεξή. Όπω κάναμε στην περίπτωση άλλων χωρών τη Κολομβία. Δεν είναι λοιπόν μια κατάσταση όπως όλα στη ζωή που είναι άσπρη μαύρη. Και τώρα να δώσω το λόγο στον πρεσβευτή της Λέγκα πέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε πρόεδρε, προεδρεύοντα στο, στη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ και μπορώ να λάβω το λόγο για την υλοποίηση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων στην Σρι Μετά από χρόνια, η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα προχώρησε στο να ε, βάλει τη χώρα μα σε μια σωστή πορεία για την καλή κυβέρνηση, την ανθρώπινα δικαιώματα, τον κράτο δικαίου, τη δικαιοσύνη, την συμφιλίωση και την οικονομική ανάπτυξη. Οι εκλογέ έγιναν τα δύο χρόνια και προετοιμάσαν τη Σριλάνκα για αυτή την παραγωγική πορεία και την οικοδόμηση ενό δημοκρατικού καθεστώτο. Η επίσκεψη παρακολούθηση, η αποστολή παρατήρηση των εκλογών με συμμετοχή βουλευτών ε, οδήγησε στην εκπόνηση σημαντική έκθεση με συστάσει που κυβέρνησε τη Σιλάνκα ήδη υλοποιεί. Όπω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γνωρίζουν, σκοπεύουμε ενεργά και με δραστήριο τρόπο να ασχοληθούμε με την υλοποίηση του συστήματο των συμβάσεων του ΟΗΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσουμε αποκλήσει και δυσκολίε στα ανθρώπινα δικαιώματα και του σχετικού τομεί, προσπαθώντα να βρούμε τι σωστέ λύσει για να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των λαών τη χώρα μα. Πρέπει να εντοπίσουμε και συγκεκριμένου τομεί όπου χρειάζεται τεχνική βοήθεια ή οικοδόμηση δυνατοτήτων σε, με αυτήν την ε, πεποίθηση ότι η Σρι Λάγκα μπορεί να εφαρμόσει το ψήφισμα 3001 με τίτλο «Η πρόοδος της Σρι Λάγκα» που ομόφωνα ε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των ε, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων φροντίζουμε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση αυτή που ονομάζεται και προδοσία ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει δράση ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατευτούν. Όπου υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπρέπεια και την των ανθρώπων, να ε, υπάρξει και ανάλογη δράση. Η κοινωνία να ενισχυθεί, να υπάρχει πίστη ε, στο δικαστικό σύστημα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του και την ανεξαρτησία όλων των ε, σχετικών κλάδων. Ε, οι μεταρρυθμίση ξεκίνησαν πριν το 2015. Χιλιάδες άφησαν την Σριλάνκα τότε ως πρόσφυγες. Ε, ε, έχουν επιστρέψει όμως και μας βοηθούν να εδραιώσουμε αυτή την διαδικασία συμφιλίωσης. Όπως προχωρούμε σε αυτό, τον, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, Χρειαζόμαστε ε, μακροπρόθεσμο βλέμμα και όχι να επικεντρωθούμε σε κοντόφθαλμα ε, πολιτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί όλη η κοινωνία ε, σε αυτέ τι προσπάθειε. Ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο ο πρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσοι επισκέφθηκαν τη και είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε όλε τι περιοχέ τη χώρα τον τελευταίο χρόνο. Οι βουλευτέ και εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση επισκέφτηκαν χωρί κανένα εμπόδιο όσε περιοχέ επιθύμησαν. Λαμβάνουμε υπόψη την έκθεση του Υπατεκούς από τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΙΕ, πολύ σοβαρά υπόψη, με την λογοδοσία και την ε, διαφάνεια και την αντικειμενικότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως θα συζητηθεί στη Γενέβη με τη συμμετοχή πολλών χωρών, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και το καθεξής. Καλωσορίζουμε τις συστάσεις αυτές από το 2015 και με την ανάλογη εντολή ε, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση και την αφοσίωσή μας να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να υπάρξει δικαιοσύνη, λογοδοσία και ανεκρατήσει τα δικαστικού κλάδου στην Σρι Λάγκα. Θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των συστάσεων και θα υποβάλουμε έκθεση για την πρόοδο του χρόνου στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπήρξε απουσία διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015, αλλά έκτοτε υπήρξαν υψηλό επίπεδο επισκέψει από τη Σριλάνκα προ τι Βρυξέλλε, όπω τόνισε ο συνάδελφο από την ΕΕΔ και αντιστρόφου, και οργανώθηκαν και δημερεί συναντήσει επίπεδο αξιωματούχων. Στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για την Διακυβέρνηση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Εμπόριο και την Οικονομική ανάπτυξη στη ΛΑΚΑ παραμένει αποφουσιωμένη, αυτέ οι συναντήσει να οργανώνονται τουλάχιστον άπαξ ετησίω, ώστε να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τι προτεραιότητε και τι ε, ε, ανησυχίε των ΜΕΝ των ΔΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει πολύτιμη κοινωνική και οικονομική βοήθεια για όλε τι προσπάθειε ανακοδόμηση στη Σρι Λάκα και το εκτιμούμε βαθιά. Η ειλικρινή αυτή δέσμευση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει ξανά την ε, ε, δέσμευση των αλληλευτικών ποσοστώσεων από τη Σρι για και την αναστολή της συμφωνίας ε, όπως είχε αποφασιστεί από πέρσι Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει με την επανεξέταση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ που θα δοθεί προ τη Σρι Λάγκα, εφόσον το εγκρίνεται. Θα πρέπει να δούμε όλα τα εμπορικά θέματα που είναι πρώτη προτεραιότητα για εσά και τη Σρι και σα προσκαλούμε και εσά, Πρόεδρε να, να επισκεφτείτε τη Σρι Λάγκα για να δείτε τη χειροπιαστή πρόοδο που έχουμε επιτελέσει στην πράξη και να μα καθοδήγησετε να φτάσουμε σε μεγαλύτερη έψη και να αγγίξουμε του εθέρε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια μεστή νοήματο πρόοδο γιατί τον επόμενο μήνα μια μεικτή αντιπροσωπεία με τη συμμετοχή του πρώτου τη χώρα θα επισκεφθεί τι Βρυξέλλε για να ε, μελετήσουμε τα θέματα οικονομική εποπτεία μαζί. Ολοκληρώνοντα, Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω ότι πραγματικά ελπίζουμε να ωφεληθούμε από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ για το σχετικό μηχανισμό η μακροοικονομική σταθερότητα που μπορεί να διαφοροποιήσει τη ε, διαδικασία εξαγωγών μας μπορεί να στηρίξει μια οικονομία που ακόμη είναι έφτραυστη και πιέζεται από υψηλά χρέη. Η ε, υποστηρίξη της υπαίθρου στην, ε, ε, στις αγροτικές περιοχές της το 80% του πληθυσμού, ιδίως στο νότο και τα ανατολικά που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, προηγουμένως, είναι ο στόχος της διαδικασίας συμφιλίωσης και σταθεροποίηση. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή αυτή από τη δεκαετία του 60 έχει παραμείνει αρκετά καθυστερημένη στην πρόοδο της στο σύστημα. Λοιπόν, ε, ε, των γενικευμένων προτιμήσεων συν θα δώσει ευκαιρίες στους ε, μικρούς γεωργούς, στις γυναίκες, όσους έχουν, είναι αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα της κοινοτροφής και της γεωργίας. Και επιβεβαιώνουμε το υψηλό επίπεδο δέσμευσης να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε στενούς διμερείς δεσμούς. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας αποτελεσματικός εταίρος στο εμπόριο, την ε, βιομηχανία, την ε, γεωργία, την κοινοτομία και την έρευνα. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Αναμφίβολα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ θα φέρει οικονομικά ωφέλη στη χώρα σας και γι' αυτό πρέπει να τηρούνται και οι δεσμεύσεις. Να δώσω το λόγο στο μόνιμο εισηγητή για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ και για την Νοτιοανατολική Ασία και μετά οι υπόλοιποι. Ε, Όποιο θέλει, α σηκώσει το καρτελάκι το οποίο θέλει να ζητήσει το λόγο και η γραμματεία θα το σημειώσει. Ο Κριστό ο εισηγητής, δεν είναι εδώ, είχε θέμα με την πτήση του. Όμως θα δώσω το λόγο σε άλλο ομιλητή που θα μας παρουσιάσει τη θέση του. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά στην παρέμβασή σας. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Κρίστοφερ, είμαι ο κύριος Κασπαρή και θα έρθει αργότερα γιατί ακυρώθηκε εκτάκτως η πτήση του σήμερα το πρωί. Ε, γι' αυτό μου έστειλε την παρέμβασή του και τη διαβάζω. Πρέπει να έχουμε υπόψη δύο πράγματα υπόψη στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Πρώτον, δεν μπορούμε να περιμένουμε από καμία χώρα να είναι τέλεια. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Καναδά και την Νορβηγία. Αν ήταν ο Καναδάς και η Νορβηγία συνομιλητέ, δεν θα είχαμε αυτό το σύστημα, θα είχαμε άλλο. Δεύτερον, πρέπει να κρατήσουμε τη συζήτηση πάντοτε στο πλαίσιο των 27 συμβάσεων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να είναι ε, αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν χρησιμοποιεί το σύστημα γενικευμένο προτιμήσεων ΣΥΝ. Να παρακολουθεί δηλαδή εκ του ΣΥΝ στην εφαρμογή των 27 συμβάσεων χρησιμοποιούνται διαφορετικά ορόσημα, διαφορετικά σημεία αναφοράς για διάφορες χώρες και ελαφρύνεται η πίεση σε αυτές τις 27 συμβάσεις και γι' αυτό δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, να μην δείχνουμε ότι δεν είναι σημαντικές για μας. Είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να το καθιστούμε σαφές. Εάν η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή, ο κανονισμός ε, προβλέπει κάποια εσωπιστοχωρήσεις και δουλειά μας είναι να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι πιστοχωρήσει αυτές να είναι μικρές. Και η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών μας έδωσε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Τώρα, για τη Σρι Λάγκα. Είναι σημαντικέ οι αλλαγέ που έχει κάνει η χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια από ε, το τέλο του εμφυλίου πολέμου. Είναι μια διαφορετική χώρα από αυτή που έχασε το σύστημα γενεκεμένων προτιμήσεων συν το 2011. Όλοι οι δείκτε αυτό μα δείχνουν και δείχνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Η σημερινή Σρι Λάγκα είναι πολύ διαφορετική από αυτή του 2011. Υπάρχει μέλημα για την ισχυρή εφαρμογή των δεμεσμεύσεων, για την τακτική και συχνή εποπτεία των ε, δράσεων, περιμένουμε από τη ε, Σρι Λάγκα να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδος, πρόοδο. Ένα ζήτημα που με ανησυχεί είναι η πρόληψη των τρομοκρατικών δράσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναφέρει ως ανησυχία της. Η είπατε η εκπρόσωπος το αναφέρει ως ανησυχία και στην έκθεση για τα βασανιστήρια και στην πρόσφατη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως Κοινοβούλιο πρέπει εμείς να πούμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος γιατί η Σρι Λάγκα είναι μέρος της Διεθνούς Σύμβασης κατά των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ε, μεταχείρισης που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλωσορίζω τα βήματα που έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο της Σρι Λάγκα για την αλλαγή Τη της σχετικής και πρέπει να προειδοποιήσω για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ε, θα πρέπει να γίνουν τα δέοντα έτσι ώστε η Σρι Λάνκα να εφαρμόζει το περιεχόμενο των συμβάσεων. Να είμαστε προσεκτικοί γιατί το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, έχει ως σκοπό να κάνει τα πράγματα καλύτερα στη Σρι Λάνκα και πρέπει να μεριμνήσουμε να μην τα κάνει χειρότερα. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Καρίμ. Να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, να ευχαριστήσω τους παριστάμενους που κόμισαν την ε, εμπειρογνωμοσύνη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας πω ότι ότι ε, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, έχω συναντηθεί επανειλημμένος δύο-τρεις φορές ε, πρόσφατα και τις τελευταίες δύο φορές που τον είδα του κατέστησα σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει πλήρως το ρόλο που του αναλογεί στην εξέταση αυτής της αίτησης χορήγησης του καθεστώτος και στην διαδικασία αυτή. Και εξού και έχουμε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα. Ακολουθώντας λοιπόν το νήμα των σκέψεων του Κρίστοφερ που εξεφράστηκαν δια του στόματος του κυρίου Κασπαρίνα να πω και εγώ ότι θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη τα κριτήρια του Κοινοβουλίου να παραμείνουν ομοιόμορφα για όλες τις χώρες, να μην υπάρχει καμία απόκληση από τα κριτήρια που εφαρμόσαμε σε περίπτωση άλλων χωρών. Τώρα, ε, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο βεβαίως καλωσορίζει την τρομακτική πρόοδο που σημείωσε η Σρι Λάνκα. Αυτό είναι σαφέστατο και ε, ε, προφανές για όλους. Καλωσορίζουμε το αίτημα της Σρι Λάνκα να υπαχθεί στο καθεστώς του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ και ε, παρά τους κινδύνους μπορούμε να, έχουμε, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο εμβάθυνσης των σχέσεών μας, σχέσεων ε από τη μία και Σρι Λάνκα από την άλλη. Κάποιες ανησυχίες παραμένουν ο Ντανιέλ Κασπαρίτης ε, ανέφερε. Μιλούμε κυρίως για την πρόληψη των τρομοκρατικών ε, πράξεων και δράσεων. Η Σρι Λάγκα έχει κάποιο περιθώριο από σήμερα μέχρι το Μάιο για να ε, φέρει περισσότερα αποτελέσματα στον τομέα αυτό της πρόληψης των τρομοκρατικών δράσεων. Και υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μίλησε σήμερα για στοιχεία εντός και εκτός χώρας που ενδεχομένως επιθυμούν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία. Και γι' αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε και να διαβεβαιώσουμε ότι η διαδικασία εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμείνει ομοιόμορφη για όλες τις χώρες. Θα ήθελα να κάνω μια επικοδομητική υπόδειξη. Πιστεύω Έχοντας συζητήσει σε βάθος με πάρα πολλά μέλη και ολοκληρώνω πρόεδρε, το λέω για να παρουσιάσω κάποιε σαφεί ενδείξει ενδείξεις στην κυβέρνηση της Σρι για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ακραδάντως ότι τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετούν την συγκεκριμένη ε, άποψη ότι έχουμε μια διαδικασία monitoring three track με τρεις δρόμου το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, το διμερές και τα Ηνωμένα Έθνη. Και θα πρέπει να έχουμε και ένα τέταρτο δρόμο που θα τον βαδίσει μόνη της η Σρι Λάνκα. Δηλαδή μια αυθεντική, μια ειλικρινή δέσμευση ότι δεν θα σταματήσει στην πρόοδο που σημείωσε, αλλά θα σημειώσει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και θα χτίσει πάνω στα επιτέματά της. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκεθ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος της συντονίστριας και γι' αυτό θα διαβάσω την παρέμβαση της. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ είναι ένα εργαλείο για την ενίσχυση ανάπτυξης για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Καταργήθηκε το καθεστώς το 2010-2011 μετά από τα ευρήματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε σχετικές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε εκθέσεις από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είχαν εντοπίσει ε, ατέλειες και ελλείψεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η χώρα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις αρχές της χρονιάς θελήσαμε να αναλύσουμε την έκθεση των ΗΕ που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και να δώσουμε στους φορείς της χώρας περισσότερο χρόνο για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για να νομοθετήσουν για την πρόληψη τρομοκρατικών δράσεων, για τη μεταρρύθμιση του, ποινικού, του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Η αξιοπιστία του προγράμματος διακυβεύεται. Από τη μία πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε την προοδευτική φύση του προγράμματος και θεωρούμε ότι το σύστημα γενικεμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, εάν το δώσουμε, θα είναι το σημείο εκκίνησης για μια πιο βαθιά σχέση, πιο έντονη σχέση με τη χώρα αυτή και θα εξετάσουμε την ε, απόφασή μας επί τη βάση των σχετικών εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών Πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας ως προοδευτική. Δεν θεωρούμε ότι το σίγμα γάμα είναι μια περίληψη συγκεκριμένων συμβάσεων. Είναι ένα πολιτικό εργαλείο για να υπάρξει πολιτική βούληση και πολιτική δέσμευση με ε, τέρους. Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και σε τέτοια θέματα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικό. Το σίγμα γάμα είναι, προσφέρει πολλές δυνατότητες στη χώρα αυτή. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά στενά και θα αξιολογήσουμε τη θέση μας πριν τη λήξη της προθεσμίας τον Απρίλιο. Εν τω μεταξύ ζητώ από τον πρέσβη της Σρι Λάνκα να μας ενημερώσει για το τι έχει γίνει με την αντικατάσταση κατάσταση των προσωρικών νομιοθετικών διατάξεων για την πρόληψη τρομοκρατικών δράσεων και για τη μεταρρύθμιση του κώδικα ποινική δικονομίας. Αλλά ήθελα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες ε, πληροφορίε για τις τελευταίες εξελίξεις, τις μεταρρυθμιστικές. Ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα πέντε ομιλητέ για δύο λεπτά ο καθένα. Η επόμενη η κυρία... Merci, merci, monsieur. Ευχαριστώ Σαρνέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Το είπαν όλοι εδώ, η Σρι Λάγκα έχει επιτελέσει πρόοδο. Και θα πρέπει και εμείς να το αναγνωρίσουμε. Είναι σημαντικό, όπως ακούστηκε, να εκφραστούν βέβαια και ανησυχίε στο κοινοβουλίο μας που είναι θεμητές. Υπήρξε μια έκθεση ανησυχητική από τον ΟΗΕ για τα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάστασή του στη χώρα και βεβαίως Υπάρχει καλή θέληση στη Σρι Λάγκα, στο επίπεδο των υποσχέσεων τουλάχιστον, ε, αλλά οι υποσχέσεις αυτές πρέπει να τηρηθούν κιόλα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, τον διάλογο με τους εκπροσώπους της Σρι που θα πρέπει να είναι ανοιχτό και επικοδομητικός, και τα βήματα πρόοδου να καταγράφονται εφόσον ε, συμβαίνουν και στην πράξη, να αναγνωρίζονται και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να πλαισιώνουμε τη Σρι Λάγκα και οπωσδήποτε να μην κλείσουμε καμία πόρτα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μινέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μιλώ εκ μέρους της Λόλα Σάντσες και μου βεβαίως και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρόκειται για ένα κείμενο της Λόλα Σάντσες λοιπόν τώρα. Έχοντας παρακολουθήσει στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σρι Λάνκα, θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο καλωσορίζει τις θετικές ενέργειες της κυβέρνησης. Όμως, και πάλι ευθυγραμμιζόμενο με αυτό και άλλους διεθνείς οργανισμούς παρατηρώ ότι λίγες απτές βελτιώσεις υπάρχουν στον τομέα αυτών και θα ήθελα να απευθύνω την εξή ερώτηση για τον βαθμό εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σρι Λάνκα. Πρώτα απ' όλα, πρώτος υπουργό της Βόρειας Επαρχίας παραπονέθηκε ότι μόλις 25% της γης ε, των Ταμίλ που δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε επιστραφεί. πώ αντιμετωπίζει το ζήτημα τη επιστροφή τη ε, δεσμευμένη ε, γης από τους Ταμίλ κατά τη διάρκεια του πολέμου και ποια πρόοδο έχει συμμετοχή. Δεύτερον, όσον αφορά τι εξαφανίσει. η τελευταία γραπτή δήλωση του διεθνούς κινήματος το οποίο καταδικάζει την ατιμορρησία την οποία υπάρχει καθώς κανείς δεν είναι υπόλογος ε, από όταν υπήρξε αυτή η δήλωση τον Αύγουστο του 2016 και δεδομένων αυτών των ανησυχιών. Τι παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε για την εφαρμογή της ε, Διεθνούς Σύμβασης ε, για την προστασία ατόμων από εξαφάνιση που κύρωσε η Σρι το 2016 τον Μάιο τρίτων δεδομένων των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Σρι στη διαδικασία της συμφιλίωσης, θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρη την πρόταση του ΙΕ να υπάρξει ένα διεθνές δικαστήριο τοπικών και διεθνών δικαστών για τα εγκλήματα πολέμου. Και η άρνηση να γίνει κάτι τέτοιο ε, νομίζω ότι de facto σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν διώξει για αντεκδικήσει ε, δεδομένου δε του ιστορικού τη χώρα με ακρότες γιατί να μην συμφωνήσουμε σε υβριδικού μηχανισμού όπω προτείνει ο Επίτροπος Άνθρωπων Δικαιωμάτων και ε, να πω και εγώ δύο λόγια δικά μου θα ήθελα να επιμείνω να δώσουμε καθεστώ ε, GSP Plus ε, στην Σεριλάνκα όταν θα είναι ασφαλή τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρακολουθούν πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σολέη. Thank you, Mr. Στο κύριε Πρόεδρε, ε, θα εκπροσωπώ την Χέντι Χάουταλα, η οποία είναι σκιώδης ε, στο θέμα αυτό. Παρόλες τις εξηγήσεις που μόλις ακούσαμε από τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν, εξακολουθούμε εμείς να ασκούμε κριτική για την επαναφορά της Ριλάνκα στο καθεστώς αυτό. Οι λόγοι απόσυρσης του καθεστώντος ήταν η παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, μεταξύ 2002 και 2011 όπως ε, ε, καθώς είχε εγκριθεί ένα ψήφισμα σχετικό τον Οκτώβριο του 2015 και δόθηκε σε Σρι Λάνκα διορία μέχρι το Μάρτιο του 2017 για να εφαρμοστούν οι συστάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα επαρκούσε να περιμένουμε μέχρι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μαρτίου και την παρουσίαση της έκθεσης από τον το για να δούμε εάν θα εφαρμοστεί τώρα το καθώς ή θα περιμέναμε για περαιτέρω βελτιώσεις. Μάλιστα, η παρουσίαση της έκθεσης ε, θα γίνει αύριο στην Γενέβη, όπως ακούσαμε, αλλά η έκθεση έχει ήδη κυκλοφορήσει και λέει πως υπάρχει αργή λειτουργία της δικαιοσύνης και δεν υπάρχει λογοδοσία για τα παρελθόντα εγκλήματα και λέμε πως θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε, κάποια, σε κάποιο εκτροχιασμό της διαδικασίας. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, το Κοινοβούλιο συνομοθέτης θα πρέπει να ενσωματώσει τα ευρήματα αυτά στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Επίση λοιπόν, επειδή θα θέλαμε να υποστηρίξουμε, και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξει η κατάργηση των δασμών για την εισαγωγή προϊόντων τη Τριλάνκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθώ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αν υπάρξει κάποιο συνδυασμό των δύο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην ε, Κομισιόν. Με ψήφισμα ή χωρίς ε, των πολιτικών ομάδων ε, στην δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου, το οποίο θα εξηγεί την κατάσταση στην Σρι Λάνκα, πώς θα παρουσιάσει, πώς θα παρακολουθεί η Κομισιόν την κατάσταση στις χώρες αυτές πέρα από τις εκθέσεις του Συμβουλίου Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εκθέσεις και εγώ θα προτιμούσα να είχαμε και έναν εκπρόσωπο των Ταμίλ ο οποίος θα μας παρουσίαζε την κατάσταση για να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε πώς θα πάει η μειονότητα, πώς θα πάνε τα παιδιά, τι γίνεται με τις γυναίκες, με τη βία κατά των γυναικών. και ποιες είναι οι προσπάθειες ε, που υπάρχουν. Ε, γνωρίζουμε και την έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι είναι πολύ αργόσυρτη η διαδικασία και πως ε, χρειάζονται βελτιώσεις. Στόχος είναι βεβαίως να στηρίξουμε την Σεριλάνκα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε το καθώς γενικευμένων προτιμήσεων στη Σρι Δεν είμαι ακόμα πεπισμένη και η ιδέα αυτού του οδικού χάρτη επίση είναι καλή να μην λέμε απλά ένα ναι ή ένα όχι αλλά να βλέπουμε τις ε, βελτιώσεις ε, και την κύρωση των 27 συμβάσεων. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία είναι ασαφή και όπως είπα θα ήθελα να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο των ε, Ταμίλ για να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ, Μάρτιν, τελευταίος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν σοβαρέ βελτιώσει στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σρι Λάνκα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Επειδή ο χρόνο πιέσει, έχω τρει ερωτήσει, δύο για τον πρέσβη και μία για την Κομισιόν. Προ τον κύριο πρέσβη πρώτα. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ένας δισταγμός για να δικαστούν ε, ένστολοι, είτε μιλάμε για στρατό είτε για αστυνομία. Είναι έλλειψη βούλησης, έλλειψη δυνατότητων ή για πολιτικούς λόγους ε, δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Η δεύτερη ερώτηση προς τον πρέσβη σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μία από τις ευκολότερες προτάσεις που κάνει ο Επίτροπος είναι στην παράγραφο 66α, όπου ο ύπατος λέει ότι η κυβέρνηση της Σρι μπορεί δημοσίως ε, και αμετάκλητα να δώσει έντολες ε, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας ότι απαγορεύονται τα βασανιστήρια και οι σεξουαλικές ε, παραβιάσεις ε, δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι μια απλή δύσκολη από την κυβέρνηση. Το σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση της Ελλάδας πριν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Και τέλος η παρακολούθηση όπως είπαμε είναι κάτι το γκρίζο, αλλά ε, αν δεν οδηγεί σε κάποιες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων δεν έχει και νόημα. Και το ιστορικό Βεβαίω ε, του καθεστώτος αυτού γενικευμένων προτιμήσεων ε, μας δείχνει ότι δεν λαμβάνουμε μέτρα. Η Σρι Λάνκα ήταν η εξαίρεση ο κανόνα. θα δεσμευτεί η Κομισιόν να αναλάβει δράση αν υπάρξουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για τους ε, δικού μας. Τρία λεπτά ο καθένας. Επιτροπή. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις που απευθύνονταν στην Επιτροπή και θα αφήσω τα υπόλοιπα στους συναδέλφους της ΕΕ και στον πρεσβευτή. Νομίζω ότι ε, έγινε μια πολύ σημαντική παρατήρηση και θέλω εδώ να μοιραστώ κάποιες από τις σκέψεις μου. Δεν είναι απλά τα θέματα αυτά. Υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες και τα διλήμματα για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, αλλά θα τα βλέπουμε και σε επίπεδο καθημερινό. Το ε, σύστημά μας δεν προσφέρει ποσοτικούς δείκτες. Θα ήταν πολύ απλό να είχαμε ένα πίνακα και να συμπληρώνουμε κουτάκια. Έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις λίγο πιο περίπλοκες. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί μια απόφαση ούτως ή άλλως. Όπω είπα προηγουμένω, δύο λόγια παραπάνω για την προσπάθεια παρακολούθηση και αποκτήρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόεδρε. Το, το είπατε κι εσεί. Η κατάσταση δεν είναι πάντοτε άσπρο ή μαύρο. Συμφωνούμε απολύτω. Η δυσκολία είναι 50 αποχρώσει στον κρύο ενδιάμεσα για να δούμε πού θα ε, μπει ο σωστό ε, ο δείκτη ακριβώ. Ως προς τους οδικούς χάρτες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τι νομικέ απαιτήσει του κανονισμού. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε του δείκτε κριτική αξιολόγηση ή τα σύνολα και τα συναθρίσματα που χρησιμοποιούμε και να ζητήσουμε τη Σελάγκα να κάνει τελείω διαφορετικά πράγματα από ό,τι ζητάμε από άλλου δικαιούχου. Επειδή όμω έχουμε το σύστημα παρακολούθηση του μηχανισμού ε, συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, θα πρέπει να δούμε εάν με κάποιο οδικό χάρτη θα βοηθήσουμε την Σελάγκα να προχωρήσει στη σωστή υλοποίηση και να τηρήσει τι δεσμεύσει τη. Ω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε ότι έχουμε κάπω διαφορετικό μηχανισμό σε σχέση με προηγούμενου κανονισμού ε, συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Έχουμε έναν αρκετά προηγούμενο τρόπο ανταλλαγή πληροφοριών με την κυβέρνηση, είτε με έναν κατάλογο που αναφέρουμε όλε τι ελλείψει και περνάμε σε συζήτηση σημείο προ το σημείο, περιμένοντα η κυβέρνηση να δώσει κάποια απάντηση. Αλλά σε αυτή την φάση σχεδιάζουμε, αν όλα πάνε καλά και η πάρει αυτό το καθεστώ ΣΥΝ, να στείλουμε ήδη μια αποστολή πολύ ε, αυτό το χρόνο, αυτή τη χρονιά κιόλα, προκειμένου να προετοιμαστεί η έκθεση. Η δεύτερη έκθεση του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να είναι έτοιμη στο τέλο τη χρονιά, όπω ξέρετε. Θέλουμε η Σρι Λάνκα να μπορέσει να αναφέρει βήματα πρόοδου σε αυτή την έκθεση, εξηγώντα βεβαίω κατά λεπτό και ελλείψει και πώ η κυβέρνηση σκοπεύει να τι αντιμετωπίσει. Πολύ σύντομα να προσθέσω ότι σε τέτοιε καταστάσει βεβαίω. Χρειάζεται μια ε, συγκεκριμένη πορεία, μια ρότα στο ταξίδι μας. Ε, η Επιτροπή θα ενημερώσει για το κατά πόσον η κυβέρνηση μπορεί να ε, ακολουθήσει την υλοποίηση του μηχανισμού συστήματος γεννηθωμένων προτιμήσεων. Ευχαριστούμε η ΕΔ. Ευχαριστώ. Για την αξιολόγηση της υπό εκπροσώπου στη Γενέβη και το κατά πόσον αυτό συμπίπτει με τη δική μας την αξιολόγηση, η απάντηση είναι ναι. Συμπίπτουν. Συμφωνούμε. Υπήρξε κατά πρόοδος, αργή όμως, και πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση και τους ε, φορείς του ΙΕ, ως προς την ατιμορρησία και τα βασανιστήρια συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο των εργασιών μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί ο Πρωθυπουργό μας έδωσε την ε, επιβεβαίωσή του ότι είναι μηδενική η ανοχή της κυβέρνησης προς τα βασανιστήρια. Και αυτό δηλώθηκε και δημοσίως από τον Υπουργό Εξωτερικών στη Γενέβη, στην σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως προς την επιστροφή των γεών εδώ ακούμε διαφορετικού αριθμού από την κυβέρνηση διαρκώ για το πώ η γη έχει επιστραφεί ποιε εκτάσει δηλαδή σε σχέση με τα όσα δηλώθηκαν εδώ, θα πρέπει να επαληθευτούν αυτά τα στοιχεία. Αλλά αυτό που ζητήσαμε από την κυβέρνηση στο επίπεδο τη ομάδα εργασία και στι συναντήσει με του πρωθυπουργού και τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράση διαφανέ με πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των γιών. Αυτό είναι αυτό που ζητήσαμε εμεί. Ευχαριστούμε και τώρα εσεί, κύριε Πεσεφτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτέ για τις ε, παρατηρήσει του. Τις ανησυχίε σα κατά μεγάλο μέρος τις συμμεριζόμαστε και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο περισσότερα μπορώ. Για τον νόμο κατά τη θερμοκρατία που πρόκειται να αναστείλει τον νόμο περί θερμοκρατία, ένα νόμο τον οποίο προωθησαν μόνο ορισμένα μονομένα άτομα, αλλά τώρα όλοι οι συνομιλητέ και ενδιαφερόμενοι έχουν συμμετάσχει στι διαβουλεύσει για την πρόθεση αυτού του νόμου. Θα ε, έχουμε έγκριση, ελπίζω σύντομα, καθώς οι Υπουργοί πέρασαν τον νόμο τον Ιανουάριο του 2017, θα υπάρξει και έγκριση από το Συμβούλιο Ασφάλειας, ένα νέο μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί για να υπάρχει συμφωνία των εταίρων, και ε, συμβουλευτήκαμε και εμπειρογνώμες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπόνηση του νόμου αυτού. Ελπίζουμε ότι η τελική έγκριση για τον νόμο θα φτάσει στα τέλη του μήνα. Για τις ποινικέ διαδικασίες η κυβέρνηση ενέκρινε την αναθεώρηση του σχετικού κώδικα που προβλέπει ότι ένας ύποπτος πρέπει να έχει και ε, υποστήριξη από συνήγορο ε, για τα θέματα των γεών τον περασμένο χρόνο Έχουμε επιστρέψει περίπου 9.000 ε, εκτάρια. 9.000 άκρα λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε ούτως ή άλλως έναν ανεξάρτητο και αντικειμενικό μηχανισμό ε, στα πλαίσια του, ε, μηχανισμού. του Τη προσπάθειε επιστροφή των γεωνών με τη συμμετοχή των γεών, με τη συμμετοχή όλων εμπειρογνωμόνων, πολιτών, ε, ε εκπροσώπων τη κυβέρνηση και ούτω καθεξή. Και αυτό γιατί δεν είχαμε έναν εξάρτητο δικαστικό σύστημα ω τώρα. Έχει επιτελεστεί πολύ πρόοδο πάντως Ελπίζουμε θα γίνουν και άλλες προσπάθειες και θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα από την πλευρά της Σρι Λάγκας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τους μας. Πρέπει να αποφασίσουμε βεβαίω από τι διαδικασίες εδώ πολύ σύντομα. Θα κλείσω τώρα τη συζήτηση για να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Και πριν περάσουμε στο σημείο 10 λοιπόν, να ελέγξουμε κατά πόσον όλοι να ακούσουμε και να, να δούμε μάλλον, ε, να δοκιμάσουμε τις κάρτες για την ψηφοφορία. I can find my voting card. Okay. Δεν βρίσκω την κάρτα μου. Καλά. So, has everybody voted? Εψήφισαν άπαντες. And the vote is closed. Πέρας. In track and we have one extra vote from... Υπάρχει ένας παραπάνω. Σημείο 10, Ταμείο Εγγύηση για την Εξωτερική Δράση. Λοιπόν, τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ αποχές κατά δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική ισοφορία άρχεται ηλεκτρονικά. Και πέρας. Και η κυρία Μπεγκίν υπέρ, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις εξωτερικές πτυχές. Εξωτερική διάσταση, όπως ε, λέμε, τη ΣΕΡΑΜ. Λοιπόν, για να μην έχουμε προβλήματα. Έχουμε την τροπολογία 40 λοιπόν πρώτη. Ποιος είναι υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Α, συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική 1 αυτή είναι η πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεκτή. Μετά περνάμε στην τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 40 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και η κυρία Μπεγκίν. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 45, κάτι το γλωσσικό, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 46, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 49 και 50 ταυτόσιμε υπέρ. Κατά. αποχέ. δεκτή. Και 51 και 51 μαζί. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν το βλέπω να το υπαλληθεύσουμε. 53 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Ε, Και η κυρία Μπεγκίν υπέρ, αλλά παρόλα αυτά απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. 68. Ε, Να δούμε και τη ψηφοφορία. Πέρας. Είδατε μάτι που έχω λοιπόν δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 79 υπέρ 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική ε, συγγνώμη τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στα εκτιμώντας Λάθος. 124. Τροπολογία 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τροπολογία 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε τροπολογία 12 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Και η κυρία Μπιγκίν τώρα έχει την κάρτα της. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Να το ξαναδούμε. 18 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβεστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 28 άρχη τη ψηφοφορία πέρας δεκτή Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Και μετά ερνάμε στην τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και περνάμε στις ε, τοποθετήσεις άλλων επιτροπών. Από την Επιτροπή Ελεγκτού του Υπερπολογισμού. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο της ελέγχου του υπερπολογισμού υπέρ κατά αποχές δεκτή. Control 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές δεκτό β υπέρ κατά αποχές δεκτό σ υπέρ κατά αποχές δεκτό ε υπέρ κατά αποχές δεκτό, F υπέρ κατά αποχές δεκτό, G υπέρ κατά αποχές δεκτό και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μπεγκίνη. Σημείο 12. Έκθεση για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας και έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά εποχές θα το επαληθεύσουμε 28 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά Αποχέ. εδεκτό Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εδεκτή Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 40 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. εδεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9, ε, τροπολογία 9, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, α, 10, 10, με συγχωρείτε, τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην νομοδότηση της ΕΜΠΛ. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Παραγραφός 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Και... Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας F Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται συγχαρητήρια. Σημείο 13 λοιπόν και εδώ να σας πω ότι οι συντονιστές χτες λόγω των α, τελευταίων εξελίξεων αποφάσισαν να αναβληθεί αυτή η και περνάμε σημείο 14 έχουμε αφενός την ε, συνένεση για την συμφωνία με Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, μία ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και αυτό με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται και... Παράλληλα με αυτό έχουμε και μια προφορική ε, ερώτηση που έχετε μπροστά σας, ε, το κείμενο το αποφάσισαν οι συντονιστές και αυτή μια ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτή την προφορική ερώτηση. Και... Πέρασε. Και αυτό με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες και περνάμε στο σημείο 15. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Δύο συνεδρίασαν. Το ένα ήταν η ομάδα παρακολούθησης ε, της Αζίαν. David, πες μας τι έγινε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Η ομάδα εποπτείας ΑΣΕΑΝ ε, των πέντε ε, ε, υπάρχει για να μην ε, α, αντιμετωπίζουμε μια χώρα σε τέτα τέτ. Για την Ινδονησία ασχολήθηκε με τρεις χώρες η ομάδα. στην Ινδονησία έγιναν δύο γύροι διαπραγματεύσουν ο τελευταίος 24 με 27 πρώτου στον Παλί. Πολύ ωραία ήταν. Οι διαπραγματεύσεις είναι βεβαίως σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μίλησαν για τους κανόνες προέλευσης για τις δημόσιες ε, συμβάσεις, για τη διανοητική ιδιοκτησία, για τον ανταγωνισμό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα γνωστά θέματα. Ωστόσο, για τις δημόσιες συμβάσεις δεν είμαστε και τόσο ενθουσιώδεις. Για το φινικέλεο η ομάδα εργασίας για το εμπόριο και τις επενδύσεις συσκέφθηκε μετά το γύρο για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και υπήρξε δέσμευση να έχουμε μέχρι το 2020 ένα σύστημα πιστοποίηση στην Ινδονησία για την ε, παραγωγή φινικελαίου με σεβασμό στα προεπαιτούμενα στο περιβάλλον και σε όλα αυτά τα οποία εμάς μας ε, ε, ενδιαφέρον. Η Ινδονησία έχει θετήσει κάποια προστατευτικά μέτρα ως προς τα γαλακτομικά μεταξύ άλλων. Τώρα για τις Φιλιππίνες έγινε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων το Φεβρουάριο για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα πολύ καλά οργανωμένη, οι τεχνικές συζητήσεις προχωρούν εξαιρετικά καλά, αλλά πρέπει κανείς να γνωρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, λαμβάνουν χώρα, διενεργούνται και την υποτισέμενη μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, κάτι που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, υπάρχει απειλή ε, για τη θέσπιση θανατικής ποινής Και έχουμε και extrajudicial killings. Η απάντηση του Προέδρου των Φιλιππινών στο, ψήφισμά μας ήταν ιδιαίτερα ε, ανησυχητική γιατί μας είπε να πάμε από εκεί που ήρθαμε και να μας ενδιαφέρει μόνο η δουλειά μας και τα δικά μας. Εμάς όμως είναι η δουλειά μας γιατί οι Φιλιππιάνες εποφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ και έχουμε δικαίωμα να το αποσύρουμε. Άρα ε, δεν έχει δίκιο ο πρόεδρος των Φιλιππινών όταν λέει ότι δεν είναι δική μας δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόθεση να προγραμματίσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων και θα περιμένουμε την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γάμα σίγμα πι Πρόσφατα υπέγραψε αυτή η χώρα τη Συμφωνία των Παρισίων και έχει ξεκινήσει εγχώρια διαδικασία κύρωσης της ε, ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τη Μιανμάρ δεν έχουμε Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου, αλλά Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων. Και Είμαστε κοντά στη σύναψη αυτής της συμφωνίας και θα έχουμε το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτών, Investment Court System, το ICS, και θα έχουμε και στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης στη συνολική συμφωνία. Είναι κάτι που δίνει ασφάλεια στους επενδυτές μας, αλλά είναι καλό και για τη Μιανμάρ, γιατί μπορούμε να εξάγουμε πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα αυτή. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο η Μιανμάρ μεταχειρίζεται τον πληθυσμό Ροχίνγκίγια. Δύσκολο να εγκρίνουμε την επενδυτική συμφωνία όταν συνεχίζονται αυτές οι καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τη Μιανμάρ και την Ινδοσία είναι καλή πρόοδος, αλλά το πολιτικό πλαίσιο και στις τρεις χώρες δεν είναι και το ιδανικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πράγματι θετικά τα τεχνικά, αλλά αρνητικά τα πολιτικά. Ας ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία. Μία δεύτερη ομάδα εποπτείας και παρακολούθησης ήταν για άλλες χώρες, για τις αφρικανικές χώρες. Είχαμε ε, τρίτη συνεδρίαση με θέμα την αηφορία. Ο κύριος Σόλτς είναι εδώ. Ε, ζητώ συγνώμη για τις χώρες των Άνδεων. Ο κύριος Σόλτς να μας ενημερώσει παρακαλώ. Πρόεδρε. Πρόεδρε, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, διότι συνδυάσαμε ακρόαση για την κατάσταση της ε, υλοποίησης, της ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και σύνδεσης με την Κολομπία, το Περού και το Εκουαδόρ. Όλα αυτά θα προσταθούν στο κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Δηλαδή τα θέματα που μας ενδιαφέρουν καλύπτονται ή τέλο πάντων προχωρούν κατά τη διάρκεια των ε, δημοτάσεων αυτών. Παρακολουθούνται και από την ΑΕΔ και την κοινωνία των πολιτών χρειάζεται μια συνοπτική εικόνα για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υλοποίηση του ε, χάρτη, μια από τις βασικές μέρημνες του Κοινοβουλίου, για τις διάφορες εις και σφαιρικές συμφωνίες. Κάποια πρόοδος έχει επιτελεστεί, αλλά από τη δική μου την άποψη ως εισηγητού, η πρόσβαση, η προσχώρηση του Εκουαδόρ δεν, θα είναι, δεν είναι ακόμα ε, σε καλή πρόοδο. Η Κολομβία σέβεται τη θέση μας, όπως εκφράστηκε από το ψήφισμα και τον οδικό χάρτη, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε τι πρόοδος μπορεί να γίνει. και θα πρέπει να επηρεάσουμε και τη δουλειά των μεικτών επιτροπών για το θέμα των συνοδευτικών μέτρων του οδικού χάρτη, ώστε να υπάρχει το σωστό follow-up. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί και μια μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς έχει προχωρήσει η υλοποίηση της συμφωνίας. ώστε να υπάρξει μια θετική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη των τριών χρόνων για τι οποίε συζητούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσει. Όχι. Και πάλι λοιπόν. Οι ομάδες αυτές θα παρακολουθήσουν την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο σημείο 16. Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος, η ΚΑΚ. Και τώρα ο εισηγητής μας, ο κύριος Γουάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για να πω ότι αυτή η Επιτροπή για το Βαμβάκι Ιδρύθηκε το 1999, είναι μια διεθνής επιτροπή των βασικών προϊόντων βάμβακος. Συμμετέχουν 27 χώρες παραγωγή και κάποιες καταναλώτριες χώρες. Είναι το μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως για τα βασικά προϊόντα βάμβακος και ασχολείται με τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων και μια διεθνή αγορά υγιή και εύρωστη για το βαμβάκι. Η Επιτροπή αυτή είναι από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς βασικών προϊόντων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει ακόμα. Παρόλο που εννέα από τα κράτη-μέλη είναι συνδεδεμένα ή συνεργάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε άλλε διεθνεί οργανώσει για ε, βασικά προϊόντα, όπω η ζάχαρη, το λάδι, ο καφέ. Οπότε δεν είναι και πολύ σαφέ γιατί δεν συμμετέσχει σε αυτό το διεθνή οργανισμό. Από το 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί την προσχώρηση σε αυτόν τον οργανισμό. Τελικά το 2013 ξεκίνησαν διαπραγματεύσει ενημερώνοντα τα εννέα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη ότι μπορούν να αποσυρθούν από τον οργανισμό για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει πλήρω εκπροσωπώντα τα η ποσότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά θα είναι μικρότερης αξίας από ότι οι εννέα ποσοστώσει των μελών που τώρα συμμετέχουν ε, συναπτυζόμενες. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον οργανισμό γιατί είναι μεγάλη σημασία του Παντακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για την οικονομία κάποιων κρατών μελών αλλά και για την βιομηχανία φαντουργικών και ένδυση ε, καθώ και άλλου εμπορικού κλάδου που ενδιαφέρουν του χονδρέμπορου και του λιανοπολιτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 6.000 παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έχουμε γίνει ε, εισαγωγική κατεύθυνση, τόπος εισαγωγών παρά εξαγωγών από το 2010. Η προηγούμενη έκθεση ήταν υπό την εποπτεία της κυρίας Μοσκαρδίνη. Είχε συσταθεί από τότε η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οργανισμό του Βάμβακος. Η βιομηχανία αυτή έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούμε εφάσματα από βαμβάκι σε μεγάλο βαθμό στην ε, Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και αυτή η πρώτη ύλη είναι ένας κλάδος ε, πολύ σημαντικός που αφορά και την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια. Και θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και την ε, αφρικανική παραγωγή προϊόντων πάμπακος. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω κάποιε ανησυχίε και προκλήσει που μα ενδιαφέρουν σε σχέση με αυτόν τον ε, τομέα. Πρώτα πρώτα, όλοι οι παράγοντε ε, του ε, κλάδου αυτού θα πρέπει να συνεργάζονται στο επίπεδο τη Επιτροπή ώστε να, αποφύ... να, αντιμετωπίσουν την υποβάθμιση των πολιτικών συνθήκων στη Μέση Ανατολή. Επίση, θα πρέπει να ελέγχονται τα εργασιακά δικαιώματα σε όλη την αλυσίδα παραγωγή προϊόντων βάμβακο. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκε ώστε η παραγωγή των αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν πρόσβαση στις βασικές αλυσίδε παραγωγής αξιών. Επίσης, η Κίνα, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός ε, βάμβακο και προϊόντων βάμπακος και ο η χώρα που έχει τη μεγαλύτερα μερίδια τη αγορά παγκοσμίω, θα πρέπει να πιεστεί για να αναλάβει σχετική δράση. Και όλε οι χώρε που ασχολούνται με το τομέα του βάμβακο να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο κλίμα για την διάδοση καλύτερων πρακτικών στα εργασιακά και την επιβολή τους κυβερνήσει, οι εκπρόσωποι εργοζομένων και εργοδοτών, οι συνδικαλιστικές οργανώσει και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τη δράση του και τη δουλειά του, προσπαθώντα να πετύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά του βάμβακο και τη ένδυσης και να υπάρχει και καλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εξάλλου, οι εξαγωγές προϊόντων βάμβακος και άλλες ε, δράσεις που θα μπορούσαν να ε, αναλυθούν ως πρωτοβουλίες μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις διακυμάνσεις των τιμών. Ε, είναι ένας ε, τομέας ο οποίος θα μπορούσε να εφεληθεί και από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά δεδομένα επίσης και η συλλογή πληροφοριών, καθώς και η παρακολούθηση των αλυσίδων, των αλυσίδων παραγωγής και προμήθειας είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να παρακολουθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν αυτό που θα είχα να στήσω εγώ στην Επιτροπή μας είναι να εγκρίνει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ε, Επιτροπή αυτή ως πλήρου μέλου. μέλους. Ε, ευχαριστούμε και τώρα λόγω στους κοιόδης εισηγητές για τους σοσιαλιστές η κυρία Χιονγκέριους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Εδώ έχουμε μια πολύ αναμενόμενη διαδικασία προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Διεθνή Επιτροπή για το Βάμβακα. Καλό θα ήταν λοιπόν να προχωρήσουμε αμελητή και με βήμα ταχύ. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε πολύ ισχυρότερη φωνή σε αυτή την Επιτροπή, γιατί υπάρχουν πολλά εναπομείναντα προβλήματα σε σχέση με την παραγωγή αυτού του σημαντικότατου ε, είδους, ε, την παιδική εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα γενικώ. Ε, αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλό θα ήταν λοιπόν οι ανησυχίε μα να ακουστούν και ενδεχομένω να ε, βρουν και τη σωστή απάντηση στο επίπεδο τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέσω των εκπροσώπων μα. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για μια βιώσιμη αλυσίδα αξιών του Βάμπακος. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν βλέπω άλλους σκιώδες εδώ. Χέλμουτ, θα την καταστήσεις στη Λόλα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ε, σκιώδους εισηγήτριας θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη συνεισφορά της και θέλω να πω ότι η χώρα μας είναι υπέρ της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός παίκτη στην παγκόσμια αγορά, αγορά υφαντουργίας. Η παραγωγή μας είναι ένα μικρό μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής. Εισάγουμε πάρα πολλά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όμως πρέπει να εμπλακούμε, να είμαστε μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας δημιουργίας αξιών, εξού και είναι ανάγκη οι δράσεις μας να παρουσιάζουν συνοχή και συνέπεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος δωρητής στον αφρικανικό τομέα βάμβακος. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα πολύ μακροσκελές βιβλίο τη σύγχρονη ιστορία του καπιταλισμού ο βασιλιάς Βαβάκη, King Cotton, από έναν καθηγητή του Χάρβαρτ. Περιγράφει την πορεία ενός προϊόντος ο Σβέν Μπέκερτ καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την κατανάλωση, την παραγωγή. Ε, τι έκαναν οι αρχαίοι παραγωγοί του βάμβακο στην Κίνα και στην Ινδία όταν ε, έχασαν αυτή την αγορά από τους Πορτογάλους και το Ηνωμένο Βασίλειο όταν έφτασαν ως νέοι απικιοκράτες στις περιοχές αυτές του κόσμου όπου κατέλαβαν την αγορά και οργάνωσαν το μοντέλο παραγωγής και εξαγωγής στην Ευρώπη. Εξαγωγή στις χώρες αυτές από την Ευρώπη λοιπόν των απεικιοκρατών. Τώρα έχει γίνει το αντίστροφο και εμείς εισάγουμε από αυτές τις περιοχές του κόσμου. Ε, κάνει μια ιστορική αναδρομή λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όλοι συμφωνούμε και θεωρούμε ότι είναι ένας κλάδος στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη, θα πρέπει να τηρούνται τα, τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά θα ενισχυθούν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή ε, Βάμβακος. Ευχαριστώ. Ποιο ήταν το όνομα του βιβλίου, ο τίτλος του βιβλίου King Cotton, απαντάει ο ομιλητής, ο βασιλιάς Βαβάκη, μια σύγχρονη ιστορία του καπιταλισμού. Δίνω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο εισηγητής, η εισηγήτρια διαμέσου του κυρίου Σόλτς, όντως είναι ο χαμένος κρίκος στην αλυσίδα των ε, βασικών προϊόντων και της διακίνησης αυτών σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στα αντίστοιχα συμβούλια για, τα, για τη ζάχαρη, για τον καφέ, Επομένως η παρουσία της ε, ε, στο Διεθνές Αυτοσυμβούλιο, σε αυτή τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή θα προσδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το απαραίτητο ειδικό βάρος ε, για να μπορέσει να βελτιώσει τα πρότυπα, τα στάνταρ, να μπορέσει να θέσει επιτάπητος θέματα αηφορίας, θέματα βοήθειας αναπτυξιακής, θέματα αηφόρου πρώτης ύλης, βιολογικής παραγωγής βάμβακος ή μη, ε, και διάφορα άλλα λεπτά ζητήματα. Άρα το θέμα είναι να τοποθετηθούμε στρατηγικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι από την συνολική παγκόσμια λυσίδα παραγωγής αξιών ε, ε, στο τομέα της βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας και βιομηχανίας Βάμβακος. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη Γενική Διεύθυνση για θέματα γεωργίας και άλλες αρμόδιες ε, υπηρεσίες. Πράγματα πράγματι δεν είναι μεγάλη παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 300.000 τόνοι. Υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες, αλλά είμαστε και βασικός παίκτη σε, στο παγκόσμιο επίπεδο. Και η παρουσία μας στο, στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα μας δώσει τη δυνατότητα μόχλευσης να παρακολουθούμε τις τιμές και να θέτουμε τα πρότυπα. Standard setting. Είναι πολύ σημαντικό. Και ε, όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Ασία αλλά και την Νότια Αμερική. Ο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Και να πω ότι και εγώ θεωρώ απαραίτητη την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την Συμβουλευτική Επιτροπή από τον Ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία για την υποβολή πολιτιών 22 Μαρτίου. 5 το απόγευμα. 5 μου μου. Μετά μεσημβρίας. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πάντως 22 Μαρτίου 5 το απόγευμα. Ψηφοφορία 3 και 4 Μαΐου. Ολοκληρώσαμε τώρα Στη συζήτησή μας για την πρωινή συνεδρίαση θα ξαναρχίσουμε στις 3.30 και κλεισμένων των θυρών. Και στις 5 θα έχουμε την ακρόασή μας για τη διπλή χρήση. Στις 11.30 θα υπάρξει και η τελετή βεβαίω για την 60η επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Ρώμης στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ.